Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν βλέπω κανέναν άρενα συνάδελφο, οπότε αγαπητές ε, συναδέλφισες, έχουμε έξι κυρίες Νομίζω ότι αρκούν αυτές για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχουμε και τον Επίτροπο. Ας ξεκινήσουμε την ε, σύνοδο. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς την έκθεση για τα νέα τρόφιμα της κυρίας Λιωτάρ. Η κυρία Λιωτάρ είναι η συγγήτρια, έχει το λόγο ε, για τέσσερα λεπτά για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Έχετε το λόγο voorzitter vriendelijk bedankt. Eh, αγαπητέ πρόεδρε σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους σκιώδεις εισηγητές, ακόμη και εκείνους που δεν είναι παρόντες για τη συνεργασία τους. Ο νέος κανονισμός για τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να διευρυνθεί για να λάβει υπόψη και τα θέματα διατροφικής ασφάλειας, γιατί τα τρόφιμα ε, παίζουν σημαντικό ρόλο για τους καταναλωτές. Ε, επίσης το περιβάλλον, τα διοντολογικά προβλήματα, η ευζοία των ζώων, όλα αυτά τα στοιχεία συνδέονται με τα τρόφιμα. Η καινοτομία καλό πράγμα είναι φυσικά, αλλά δεν θα πρέπει να είναι επιζήμια για την υγεία την ποιότητα ζωής ε, των ατόμων. Ελπίζω ότι οι περισσότεροι βουλευτές θα συμφωνήσουν με αυτές τις ιδέες που σας διατυπώνω. Τι εννοούμε με τον όρο νέα τρόφιμα. Είναι προϊόντα τα οποία δεν υπήρχαν στην αγορά, την ευρωπαϊκή αγορά, πριν από τις 15 Μαΐου του 1995, γιατί δεν είχαν ε, επινοηθεί ή γιατί δεν είχαν τεθεί σε εμπορία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα παράδειγμα των νέων τεχνολογιών που υπάρχουν πια στην αγορά. Τώρα για τον καταναλωτή οι καινοτομίε είναι πάντα ενδιαφέρουσε. και οι τεχνολογίες θα μπορούσαν να μα ε, βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε α πούμε την παχυσαρκία. Αλλά πρέπει να είμαστε συνετοί και προσεκτικοί ε, σε ό,τι αφορά τη θέση σε... στην αγορά προϊόντων ε, όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι επιζήμια, ότι είναι επωφελή για την υγεία. μπορεί να υπάρχει κάποια υπόνοια ότι είναι επιβλαβή για την υγεία. Επίση, για τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να ισχύει η αρχή τη ε, προφύλαξη. Ε, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εγγύηση. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλή. Θα πρέπει βέβαια οι καταναλωτέ να έχουν τη, δυνατότητα επιλογή για όλα τα τρόφιμα και για τα νέα τρόφιμα και αυτό προποθέτει καλή ετικετοθοσία. Ε, τα τρόφιμα τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή από τους ε, απογόνους τους μας δημιουργούν ένα επιπλέον πρόβλημα είναι προϊόντα τα οποία ε, είναι αποτέλεσμα δοκιμών που έγιναν ε, λαμβάνοντας υπόψη ή όχι την ε, ευζοία των ζώων. Θα πρέπει εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστήσουμε προτεραιότητά μας αυτή την ευζοία των ζώων. Τα κλωνοποιημένα ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να τεθούν στην αγορά. Δεν είναι σωστή εμπορική πρακτική, αλλά στο μέλλον μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κρέας κλωνοποιημένων ζώων ή των απογόνων τους συζήτηση για το κρέας αυτό δεν είναι καινούρια. Το 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε την κλωνοποίηση των ζώων. Το 2008 υιοθετήθηκε ένα ψήφισμα για την εμπορία του, του κρέατος αυτού από κλωνοποιημένα ζώα ε, για να υπάρξει ένα πλαίσιο νομοθετικό. Και σε συμφωνία με το Συμβούλιο λέμε ότι τα ζώα και το κρέας των κλωνοποιημένων ζώων ε, θα πρέπει να καλύπτεται από τη νέα νομοθεσία για τα τρόφιμα. Στη δεύτερη ανάγνωση το Κοινοβούλιο όμως δεν συμφώνησε με το Συμβούλιο. Εάν, ε, για να συμφωνήσει μάλλον το Κοινοβούλιο με την ε, εισαγωγή αυτού του κλωνοποιημένου κρέατος στην νομοθεσία ε, φοβάμαι ότι θα βρεθούμε σε μια κατάσταση πάρα πολύ λεπτή. Επίσης, η νέα νομοθεσία για τα τρόφιμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ασφαλή κατανάλωση. Αλλά από την άλλη δεν ασχολείται πολύ με την ευζόγεια των ζώων και με το περιβάλλον. Μήπως θα πρέπει να έχουμε ειδική νομοθεσία για τα κλωνοποιημένα ζώα και το κρέας των κλωνοποιημένων ζώων και μήπως έτσι θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα. Πριν από λίγου μήνε αποφασίσαμε την εμπορευματοποίηση αυτών των προϊόντων, αλλά χωρί αυστηρή νομοθεσία υπάρχει κίνδυνο να εμφανιστούν στι αγορέ Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια κρέατα. Ε, ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παραμείνει στη θέση του όπω έκανε τα τρία τελευταία χρόνια. Δεν θα πρέπει τελευταία στιγμή, στο παραπέντε, να βρεθούμε ενώπιον κακών εκπλήξεων. Γιατί αυτό θα αποδείκνει ότι δεν είμαστε στο ύψος των προσδοκιών των εκλογέων μας και των πολιτών μας ε, οι οποίοι θα βρεθούν ε, με κλωνοποιημένο κρέας στο πιάτο τους. Κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό. Να, Σας ευχαριστούμε επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, συνάδελφε. Θα ήθελα να σας πω ότι ω εισηγήτρια έχετε τέσσερα λεπτά στην αρχή τη συζήτηση και δύο λεπτά στο τέλο τη συζήτηση. Και υπάρχουν συνάδελφοι που προτιμούν να, να μιλήσουν και για τα έξι τους λεπτά ε, στην αρχή και στο τέλος μόνο έχουν ε, λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, εσείς ακολουθήσατε τον κανόνα, κρατήσατε το όριο των τεσσάρων λεπτών, άρα θα έχετε και δύο λεπτά στο τέλος. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο ε, Τζον Ντάλι για να τοποθετηθεί. Ε, στη, όσον αφορά ε, την ε, παρουσίαση της εισηγήτριας. Έχετε το λόγο, Επίτροπε. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, το Μάρτιο του περασμένου έτους το Κοινοβούλιο ψήφισε την πρώτη, πρώτη ανάγνωση την πρόταση για τα νέα τρόφιμα. Πολλές από τις τροπολογίες που πέρασαν ε, ενσωματώθηκαν στην ε, θέση του Συμβουλίου που υιοθετήθηκε στην πρώτη ανάγνωση το Μάρτιο αυτού του χρόνου. Η θέση του Συμβουλίου διατηρεί την αρχή της ανάγκης ε, ε, ε προηγούμενης έγκρισης για τα νέα τρόφιμα για να εξασφαλιστούν οι καταναλωτές για το γεγονός ότι οι νέες τεχνικές παραγωγής δεν, δεν εγκυμονούν κινδύνους και για τους ανθρώπους και για τα ζώα και για το περιβάλλον. Ε, η προτινόμενη πρόταση θα ε, ε, συντονίσει και θα επιταχύνει τη διαδικασία με βάση μια κεντρική αξιολόγηση από την ΕΦΣΑ και θα καθοριστούν συγκεκριμένε ημερομηνίε και χρονοδιαγράμματα σε κάθε στάδιο. Συμπεριλαμβάνεται επίση και μια βελτιωμένη αξιολόγηση τη ασφάλεια έτσι ώστε να μπορούν παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτε χώρε να εισέρχονται πιο εύκολα στην αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι για την ευρία στήριξη του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη βελτιωμένη πρόταση για την διαδικασία έγκριση. Όσον αφορά τα νάνο τονίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ε, το αίτημα για συστηματική ετικετοθεσία ε, όλων των τροφίμων που, περιέχουν, που περιλαμβάνουν νάνο Βλέπουμε λοιπόν θετικά αυτό το αίτημα. Ε, στην τέταρτη έκδοση του ε, του κειμένου θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία όσον αφορά την προσαρμογή με τι νέε συνθήκε με τις νέες διατάξεις συνθήκης Λισαβόνας, ιδιαίτερα όσον αφορά την απαραίτητη προσαρμογή ε, του ορισμού των νάνο υλικών. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια ισόρροπη λύση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η εξέταση αυτή. Όσον αφορά την κλωνοποίηση των ζώων, συμφωνώ με το Κοινοβούλιο στο ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα. Όπω θα θυμάστε, έχω αναλάβει τη δέσμευση ε, για να υποβάλουμε έκθεση όσον αφορά όλε τι πτυχέ τη κλωνοποίηση για παραγωγή τροφίμων μέχρι τον Νοέμβριο του 2010. Και στη συνέχεια θα, υπάρξουν νομοθετικέ προτάσει κατά περίπτωση. Ε, αναλαμβάνω τη δέσμευση να εξετάσουμε όλα τα ζητήματα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ε, την υγεία και την καλή διαβίωση των κλωνοποιημένων ζώων καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του, αλλά και κατά τη διάρκεια τη αναπαραγωγή η επίπτωση ε, της κλωνοποίησης στο διεθνές εμπόριο αποτελεί μια άλλη σημαντική πτυχή που θα ε, εξεταστεί στην εν λόγω έκθεση. Ε, θα, δω, θα εξετάσουμε λοιπόν τα συμπεράσματα τη έκθεση αυτή με ανοιχτό πνεύμα, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική και ισορροπημένη λύση που να μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο. Η έκθεση θα αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω συζητήσει με το στόχο να υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα για όλα τα όργανα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Λίοταρτ ε, και του όλους εισηγητέ για την πολύτιμη εργασία του ε, για το θέμα αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, τώρα περιμένω με υπομονησία να ακούσω τις απόψει των μελών του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Πίτροπε, και τώρα να δώσουμε το λόγο στα μέλη του Κοινοβουλίου, που θα τοποθετηθούν εξ ονόματος των κοινοβουλευτικών ομάδων με μεγάλη ε, χαρά να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στην κυρία Πιλάρα Γιούσο, η οποία ε, είναι συνάδελφος αλλά και συμπατριώτησα μάλιστα ε, προερχόμαστε από την ίδια περιφέρεια ε, ε, από την οποία εκλέγομαι και εγώ 22 χρόνια στο Κοινοβούλιο. Δεν είμαστε στο ίδιο κόμμα, αλλά είμαστε συμπατριώτε κυρία Γιούσο. Χαίρομαι ιδιαίτερα και σα δίνω το λόγο για δύο λεπτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για μένα αποτελεί ε, χαρά και τιμή να, το γεγονό ότι προεδρεύεται σε αυτή τη συνεδρίαση. Κύριε Επίτροπε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, όπω και εσεί είπατε, όχι μόνο για του καταναλωτέ, αλλά και για τη βιομηχανία τροφίμων. Πρόκειται για τα νέα τρόφιμα και για τι νέε διαδικασίε παραγωγή τροφίμων. Όπως ε, ε, αναφέρθηκε εδώ, ε, το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι το ζήτημα του κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα και από τους απογόνους τους. Γιατί οι απόγονοι, αν θέλετε, εντάσσονται στην αλυσίδα των τροφίμων και όχι τα κλωνοποιημένα ζώα. Ε, λοιπόν, ε, το θέμα, λοιπόν ε, το, το θέμα αυτό πραγματικά δεν δε θα μπορούσε να λυθεί μόνο μέσα από ορισμένους παραγράφους. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα καινοτόμο τεχνική, όπως αυτή της κλωνοποίησης των ζώων, παρόλο που ήδη αποτελεί συνήθεια σε ορισμένες, και ρουτίνα σε ορισμένα κράτη-μέλη. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια τροπολογία με βάση την οποία ε, ζητάμε από την Επιτροπή, όπω και εσεί υποσχεθήκατε, να υποβάλει έκθεση και νομοθετική πρόταση προ την κατεύθυνση αυτή. Εδώ λοιπόν ε, γίνεται συζήτηση και υπάρχει μια μικρή διαφωνία ακόμα και μέσα στην ομάδα μα. Αν πούμε από την Επιτροπή να ε, υποβάλει την πρόταση απαγορεύοντα. τι να πούμε, να πούμε από την Επιτροπή να απαγορεύσει την χρήση του κρέατο από κλωμμένα ζώα ή να, παρουσιά, να υποβάλει πρόταση. κατά την άποψή μου, το δεν πρέπει να ισχύσει. Δεν πρέπει εμεί να υπαγορεύσουμε στην Επιτροπή προς ποια κατεύθυνση ε, θα, θα κινείται η πρότασή της. Να υποβάλει την πρότασή της Επιτροπή και εμείς θα πούμε κατά πόσο συμφωνούμε ή όχι και θα υπάρξει τροπολογία. Ε, αυτή είναι η δική μου θέση προσωπική, αλλά είμαστε διχασμένοι στην ομάδα μας και αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε χωριστά. Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, το θέμα των υλικών. Βεβαίω, ε, απαιτείται ένα νέο ορισμό. Αλλά κοιτάξτε, τα νανοηλικά ε, δεν έχουν να, ε, ε, για, να, για να επιτρέπονται, ε, δεν πρέπει, ε, δεν αρκεί ο ορισμό ή η ετικετοθεσία. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για νέα υλικά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα τρόφιμα. Άρα λοιπόν έχει προτεραιότητα η ασφάλεια και θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένε μελέτε. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και σα ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ευχαριστούμε κυρία Αγιούσα κυρία ε, κύριε Γιούσο, ξέχασα να πω ότι μιλάτε εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ε, να το πω τώρα λοιπόν, ε, για λόγους τάξης. Τρία, λεπτά τώρα έχει στη διάθεσή της η κυρία Σάρμπου, η οποία θα τοποθετηθεί εξ ονόματος της ομάδας των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της και για τη συνεργασία με την ομάδα μας. Κύριο μέλημά μας ήταν πάντοτε η αντιμετώπιση των τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και οι επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, στην υγεία του καταναλωτή. Δεν υπάρχει επαρκή γνώση από τη χρήση αυτών των ε, τροφίμων, προερχόμενων δηλαδή από κλωνοποιημένα ζώα, ώστε να γνωρίζουμε εάν είναι ασφαλή για τους καταναλωτές ή τι είδους επιπτώσεις μπορούν να έχουν στη δημόσια υγεία όπως επίσης και προβλήματα σχετικά με την ευεξία των ζώων. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι δεν αιτιολογείται η χρήση κλωνοποιημένων προϊόντων ζώων. Επίσης, εξετάζεται το ζήτημα των νανοηλικών σε τρόφιμα ή τροφίμων που παράγονται με την νανοτεχνολογία. Δεν είναι γνωστό τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό τα νανοηλικά αυτά. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε πολύ προσεκτικοί ω προ την κατανάλωση τέτοιου είδου τροφίμων. Γι' αυτό ζητούμε ειδικέ μεθόδου αξιολόγηση από την ΕΦΣΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλεια Τροφίμων, πριν από τη διάθεση στην αγορά τέτοιου είδου τροφίμων. Πρέπει να έχουμε όσο δυνατόν πιο προσεκτική προσέγγιση σε τέτοια τεχνολογία παραγωγή νέων μορφών τροφίμων, όσο δεν γνωρίζουμε τι είδου επιπτώσει μπορεί να έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον. Επίση, πρέπει ο καταναλωτή να έχει επαρκή ενημέρωση για το τι καταναλώνει. Γι' αυτό απαιτείται να έχουμε πληρέστατη σήμανση των προϊόντων αυτών. Αποτέλεσμα της νομοθεσία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ασφαλή για τη δημόσια υγεία προϊόντα και η διαφύλαξη της ευημερία των ζώων. Υποστηρίζω κάθε λοιπόν τροπολογία που προάγει αυτούς τους δύο στόχους και τις εναλλακτικές μεθόδους για, την, ε, για τις δοκιμές τέτοιου είδους τροφίμων και μέτρηση των αποτελεσμάτων τους, έτσι ώστε να αποτρέπεται, να αποφεύγεται η χρήση τους σε πειράματα πάνω σε ζώα. Έχει προχωρήσει σε πρώτη ανάγνωση με ευρύτατη πλειοψηφία αυτή η έκθεση. Δυστυχώς όμως το Συμβούλιο δεν δέχθηκε να συμβαστεί σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κλωνοποιημένα ε, τρόφιμα προχώμενα από κλωνοποιημένα ζώα και γι' αυτό πρέπει τώρα το Κοινοβούλιο να ε, δράσει αποφασιστικά και να διαφυλάξει τα συμφέροντα των καταναλωτών. Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ. Από τους φιλελεύθερους για δύο λεπτά η κυρία Παραβάνοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία εισηγήτρια και εκ μέρους της κοιόδους εισηγήτριας μας θα ήθελα να υποστηρίξω τα, τα βασικά στοιχεία της έκθεσης που υιοθετήθηκαν και στην Επιτροπή. Όπως είπε η συνάδελφός μου, ε, τα βασικά θέματα είναι η κλωνοποίηση των ζώων, ε, τα θέματα ασφάλειας δεν έχουν ε, εντοπιστεί, για τρόφιμα τα οποία παράγονται από νανοτεχνολογία. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν προβλήματα με την βιοπικιλότητα, για την υγεία. Υπάρχουν και θέματα βεβαίω ε, διοντολογικά. Γι' αυτό θέλουμε να εξαιρέσουμε το κρέα που παράγεται από κλωνοποιημένα ζώα και του απογόνου του και ζητούμε από την Κομισιόν να παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση που να καλύπτει όλα αυτά τα στοιχεία, όλε αυτέ τι πτυχέ. Είναι απαράδεκτο να ε, ξεκινήσουμε μια διαδικασία αδειοδότηση ε, τέτοιων προϊόντων χωρί να δώσουμε την ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στου Ευρωπαίου Πολίτε τη δυνατότητα να κάνουν μια σωστή συζήτηση για τι επιπτώσει αυτή τη τεχνολογία. Και να σα υπενθυμίσω ότι αυτή τη θέση την έχουμε εκφράσει σαφώ ω Κοινοβούλιο στο ψήφισμά μα το 2008 για την κλωνοποίηση των ζώων για την αλυσίδα των τροφίμων. Σε ό,τι αφορά τα νοοτρόφιμα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι κανένα προϊόν που περιέχει σωματίδια νανοτεχνολογίας δεν θα πρέπει να τεθεί στην αγορά χωρί να υπάρχουν μέθοδοι αξιολόγηση του κινδύνου. Θα πρέπει η ΕΦΣΑ να εκπονήσει κατευθυντήριε γραμμέ ε, σε διαβούλευση με όλου του ενδιαφερόμενους κατόπιν εγκρίσεω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Θα πρέπει να συμφωνήσετε ότι το θέμα τη διαφάνεια είναι πολύ σημαντικό για αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να υπάρχει δημόσια πρόσβαση στα δεδομένα πάνω στα οποία βασίζουμε την αξιολόγηση. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δημοσιοποίηση και όλα τα δεδομένα για την αξιολόγηση κινδύνου με βάση τη σύμβαση και το ευρωπαϊκό δίκαιο να, να διασφαλίζονται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ε, με θέματα δημοσιοποίησης και δικαιώματα πνευματικά. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όταν μιλάμε επίσης για την ετικετοθεσία προϊόντων και τροφίμων που παράγονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει ένα σαφές κείμενο ε, που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στους πολίτες. Ευχαριστώ και τώρα εξ ονόματος των Πρασίνων για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Στάς. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, το 1999 όταν πρωτοεκλέχθηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έλαβα για πρώτη φορά μέρος σε συζήτηση και αυτή η συζήτηση ήταν η σχετική με την ασφάλεια των τροφίμων. Είχαμε μόλις διέλθει από το Βέλγιο την κρίση των ε, μολυσμένων με διοξίνες πουλερικών που είχε προκαλέσει τεράστιες ζημιές και είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχεθεί μια λευκή βίβλο με ε, πολύ άριθμα μέτρα για την, για, για την προστασία των ε, καταναλωτών με ασφαλή τρόφιμα. Έχουν περάσει δέκα και πάνω χρόνια έκτοτε. Πολλά έχουν γίνει. Πολύ μεγάλο μέρος της δουλειά που υποσχεθεί Επιτροπή, η Επιτροπή έχει προχωρήσει και πάνω απ' όλα βλέπουμε ότι η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να εξετάσει το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοιου είδους νέα τρόφιμα. Αυτό είναι η δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Τα νέα τρόφιμα παράγονται με τεχνολογίες που δεν ήταν διαθέσιμες πριν τις 15 Μαΐου του 1997. Η πρόταση του Ιανουαρίου του 2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε στόχο να εξυπηρετήσει μια σειρά στόχων για την ασφάλεια των τροφίμων, τη δημόσια υγεία και ε, επαρκή προμήθεια της ε, αγοράς. Η κυρία Λιωτάρ ε, ανέλαβε μια έκθεση πολύ σημαντική. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις προσπάθειές της. Καταβάλατε πολλές προσπάθειες και σε συνεργασία με μας βοηθήσατε, όπως και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορέσαμε να φτάσουμε στην πρώτη ανάγνωση σε πολύ ισχυρή πλειοψηφία υπέρ των προτάσεών σας, κυρία, κυρία Λεωνάρ μια συμπληκτική πλειοψηφία που τάχθηκε με το πλευρό σα. 658 ήταν οι βουλευτέ οι οποίοι ψήφισαν υπέρ των θέσεων σα Δυστυχώ όμω και μια και δεν έχουμε εδώ παρόντας εκπροσώπου του Συμβουλίου, καλό θα είναι να γνωρίζει το Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο μιλάει με μια ενωμένη φωνή. Προϊόντα προερχόμενα από κλωνοποιημένα ε, ζώα ή απογόνους αυτών δεν μπορούν να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Και κύριε Επίτροπε, περιμένουμε νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το χειτερό δυνατό. Εμείς οι πράσινοι θέλουμε να προχωρήσουμε ταχύτατα σε ένα μορατόριο έναντι τέτοιου είδους, τέτοιων ε, ειδών τροφίμων. Θέλουμε μια νομοθετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό και επιμένουμε σε αυτόν σε αυτή την απέτηση πρέπει η Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν να καταθέσει νομοθετική πρόταση. Πολλέ είναι τροπολογίε που υπευλήθησαν ύστερα από την πρώτη ανάγνωση. Το ΔΕ Συμβούλιο ε, επεξεργάστηκε πολύ βιαστικά και πρόχειρα την υπόθεση αυτή, δυστυχώς. Αγνόησε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων, μηνών, τις απειράριθμες συνεδριάσεις που έλαβαν ε, χώρα και δεν επέτρεψε πρόοδο στην υπόθεση αυτή. Είναι λυπηρό λοιπόν αυτό το φαινόμενο. Ελπίζω ότι στην δεύτερη ανάγνωση θα διαφυλάξουμε το ενωμένο μέτωπο, που είχαμε στην πρώτη ανάγνωση. Ίσως να χρειαστεί να φτάσουμε στην ε, συνδιαλλαγή. Εγώ συγχαίρω την κυρία Λιωτάρ για την προσέγγισή της. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ που σας δείξατε διάθεση να δεχθείτε την επανεγραφή πολλών από τις τροπολογίες που είχαμε στην πρώτη ανάγνωση, ειδικά αυτές που είχαν να κάνουν με τα κλωνοποιημένα ζώα και ελπίζω ότι μετά την ψηφοφορία το μήνυμα που θα λάβει το Συμβούλιο θα είναι απερίφραστο και σαφές. Και ελπίζω ότι θα έχουμε πλέον την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε ε, διαπραγματεύσεις ξεκάθαρες και έντιμες με το Συμβούλιο. Ελπίζω δε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει έχετε τη νομοθετική πρόταση, την οποία άλλωστε επιθυμούν όλοι οι πολίτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την ομάδα των Ελευθεριών και τη Δημοκρατία Για μισό λεπτό το λόγο έχει η κυρία Ρόσπαχ. Ευχαριστώ καταρχά την κυρία Λεωτάρη για τη δουλειά που έχει κάνει. Προσωπικώ θα ήθελα να προσπιστώ ιδιαίτερο στο δικαίωμα ενημέρωση του καταναλωτή. Αυτό ισχύει για κάθε είδο τροφίμου φυσικά. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει διάφορα στοιχεία για τις αρωματικές ουσίες ε, και λοιπά πρόσθετα που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των νανοηλικών. Πρέπει να γνωρίζουμε αν μπορεί να έχουν επίδραση στον, στην υγεία μας. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει θα πρέπει μόνο μέσα από ιατρικές διαδικασίες και με ιατρική παρακολούθηση να χρησιμοποιούνται αυτά τα τρόφιμα. Ε, περαιτέρω όμως έχουμε και το ζήτημα των κλωνοποιημένων προϊόντων, των προϊόντων από ζώα που έχουν κλωνοποιηθεί που κυκλοφορούν σε πολλέ άλλε χώρε. Και διερωτώ με ποιο είναι αυτό ο οποίο προωθεί τέτοια προϊόντα. Η βιομηχανία, η οποία απλώ θέλει να ρευστοποιήσει αυτά τα προϊόντα, να τα πουλήσει ή οι καταναλωτέ. Είναι δυνατόν ο καταναλωτή να θέλει προϊόντα στο σούπερ μάρκετ του τα οποία είναι κάπω παράξενα, τα οποία δεν είναι φυσιολογικά προϊόντα. Ε, μάλλον θέλει να έχει απλά και φυσικά προϊόντα ο καταναλωτή. Άλλωστε, βλέπουμε πόσο μεγάλη προτίμηση δείχνουν οι καταναλωτέ στα βιολογικά προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερα πρέπει να μεριμνήσουμε να ε, πολλούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα, καθαρά προϊόντα τα οποία να μην προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Στην πατρίδα μου παράγονται πάνω από 25 εκατομμύρια χείρου, ε, χείριου κρέατος ε, το χρόνο και πάνω από ένα εκατομμύριο πουλερικών χωρίς να χρειάζεται να τα κλωνοποιούμε. Ευχαριστώ. Τελειώνει λοιπόν αυτό ο κύριο παρεμβάσεων με ε, την παρέμβαση Τανασέσκου εξ ονόματο των μη διαγραμμένων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα τρόφιμα τα οποία προέρχονται από την νανοτεχνολογία πρέπει ε, να αξιολογούνται ως προς τον κίνδυνό τους πριν τους δοθεί έγκριση ε, για κυκλοφορία στην αγορά. Καθώς επίσης και τα τρόφιμα τα οποία προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους. Αυτός ο κανονισμός εξετάζει ε, το ζήτημα ε, υπό κάτω από τη σκοπιά της προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Ο όρος νέα τρόφιμα ε, φαίνεται ενδιαφέρον και μας δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για καινούργια τρόφιμα με ωραία χρώματα κτλ. Όμως η εικόνα είναι διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και βεβαίως ε, είναι θεμητή η επιθυμία αυτή για την χρήση των τροφίμων που, είναι, που προέρχονται από την ανατεχνολογία χωρίς έγκριση μπορεί πράγματι να φαίνονται ως ε, μία λύση στο πρόβλημα της πείνας κτλ. Αλλά κοιτάξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το ζήτημα της ασφάλειας και της δικής μας αλλά και των ε, επόμενων γενιών. Μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι μιλάμε για τα νέα τρόφιμα και για τα κλανοποιημένα ζώα ε, σαν κάτι το οποίο είναι το δεδομένο και, ε, και δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Να σας υποθυμίσω όμως ότι η τεχνολογία βρίσκεται σε πολλά σημεία ε, στο, σε πειραματικό στάδιο ακόμα. Και σε τελευταία ανάλυση, το ερώτημα ανάγεται στο εξή. Θα, θα δίνετε τρόφιμα αυτά στα παιδιά σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τελειώσαμε τώρα με του ομιλητέ ε, εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων και να προχωρήσουμε τώρα στη συζήτηση των συναδέλφων ε, και των επιμέρους τοποθετήσεων. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Πίτερ Λίζε για δύο λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα και εγώ προσωπικώ να εκφράσω τι ευχαριστίε μου προ την κυρία Λιωτάρ. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο μπορεί να σα υποστηρίξει ω προ τα θέματα που αφορούν τι πρόσθετε ουσίε, τα ε, τρόφιμα που έχουν ε, να κάνουν. Ε, με τις προτάσεις εμείς έχουμε διαφορετική θέση αλλά μπορούμε να βρούμε πιστεύω τη λύση. Η κυρία Πιλάρα Γιούσο έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στην συζήτηση ε, και ιδιαίτερα στο αμφιλεγόμενο θέμα των κλωνοποιημένων ζώων. Εγώ συντονιστής εκ μέρους της ομάδας μου πρέπει να σας πω ότι η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι υπέρ της απαγορεύσεως των τροφίμων και θα υπερψηφίσει αυτές τις θέσεις αύριο στην ψηφοφορία παρά το γεγονός ότι κάποιοι από την ομάδα μου ε, διαφοροποιούνται. Η συζήτηση ήταν πολύ σημαντική. Ιδιαίτερα η ειδικοί από πλευράς γεωργίας θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να διατηθένται κλωνοποιημένα ε, τρόφιμα, τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δεοντολογικές επίσης επιφυλάξεις προς την υπόθεση αυτή, αλλά πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο καταναλωτής στάστε κατά των προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Είναι τόσο πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση αυτή που είναι σαφές πως είναι αιτιολογημένη η επιφυλακτικότητα και η δυσπιστία που αισθάνεται κανείς αυθόρμητα στην υπόθεση αυτή. Είναι γνωστό ήδη ότι υποφέρουν τα κλωνοποιημένα ζώα. Ένα τρίτο εξ αυτών ε, πεθαίνει αμέσως και πολλά είναι αυτά τα οποία ε, μπορούν να επιβιώσουν μόνο μερικές εβδομάδες στην κοίηση ακόμα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι πρέπει η οποιαδήποτε νομοθεσία εισάγουμε να προστατεύει και την ευημερία των ζώων και γι' αυτό το λόγο υποστηρίζουμε τις τροπολογίες και αύριο στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιολάιναν τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπουμε ότι η κατάσταση στι πολιτικέ ομάδε παρουσιάζεται κατά τον ίδιο τρόπο και εμεί είχαμε πολύ έντονε συζητήσει, διαφοροποίηση ορισμένων ω προ τον κανονισμό αυτών. Πάντως η ευρύτατη πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ των θέσεων τη ε, εισηγήτρια και θα απευθύνουμε με τον τρόπο αυτό πιστεύω να σαφέσα το μήνυμα προ την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Νομίζω ότι συμφωνούμε κύριε Επίτροπε γιατί το είπατε και εσείς ότι στα νέα τρόφιμα υπάρχει ανάγκη να έχουμε προηγούμενη αδειοδότηση πριν από τη διάθεσή του στην αγορά δηλαδή. Και έτσι καλό θα ήταν να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα αδειοδότησης, όχι 27 διαφορετικά συστήματα αδειοδότησης από ένα, για κάθε κράτος μέλος δηλαδή, δηλαδή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις και να υπάρχει η ίδια προστασία της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων. Οι νέε τεχνολογίε μπορεί να έχουν μπει πλέον και στον χώρο των τροφίμων. Έχουμε την ανοτεχνολογία, τα νανοσωματίδια και αυτό επιτάσσει τη μέγιστη επιφυλακτικότητα και προσοχή. Όταν δεν γνωρίζουμε ακόμη τι είδου επιπτώσεις μπορεί να έχουν για τον άνθρωπο, τα τρόφιμα αυτά δεν μπορούμε να τα διαθέτουμε στα ε, καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ. Μόνο όταν θα γνωρίζουμε ότι είναι απολύτω ακίνδυνα για τον καταναλωτή μπορούμε να τα διαθέσουμε. Βεβαίως θέλουμε να έχει ο καταναλωτής και τη δυνατότητα της επιλογής. Άρα, όταν και εφόσον ε, διαδιοδοτηθούν τα προϊόντα αυτά, θέλουμε να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στη συσκευασία τους. Καλό θα ήταν την επόμενη εβδομάδα να καταλήξουμε και σε μία ε, σε μια κοινή διατύπωση, ένα κοινό ορισμό δηλαδή των ανοηλικών και να καταλήξουμε και στον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε τα θέματα της νανοτεχνολογίας. για τα κλωνοποιημένα προϊόντα από κλωνοποιημένα τρόφιμα. Ίσως θα ήταν καλό να βγει το κομμάτι αυτό, κύριε Επίτροπε, από την ε, πρόταση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να λυθούν τα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία δεν είναι αμφιλεγόμενα, κατά τρόπο απρόσκοπτο και στη συνέχεια να προκύψει νέα νομοθετική πρόταση για τα προϊόντα από κλωνοποιημένα τρόφιμα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριος Ρώση. Ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα ε, μιλάει για την αδειοδότηση των τροφίμων αυτών που μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτά τα τρόφιμα θα πρέπει να, είναι σύμμορφα με τις αρχές της ασφάλειας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θεωρούμε ότι είναι θετική η πρόταση να υποστούν αυτά τα τρόφιμα α, προληπτικούς κανόνες, ούτως ώστε να μην βάζουμε στην αγορά ε, τρόφιμα τα οποία προέρχονται από είδη τα οποία είναι παπιλούμενα. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο ε, ε, και, την εξαίρεση των τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα. Δεν συμφωνήσαμε στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά θα πρέπει η Κομισιόν να κάνει προτάσεις για την ετικετοθεσία και για την ιχνηλασιμότητα αυτού του κρέατος. Ε, θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι θέλουμε προϊόντα ε, ποιοτικά και ασφαλή. Τώρα, η κυρία Μορβάη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρόφιμα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υφίστανται ενδελεχείς ελέγχους, πράγμα το οποίο ακόμη δυστυχώς δεν έχουμε επιτύχει. Γιατί θα έπρεπε να είναι δυνατό να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο τα τρόφιμα εκείνα των οποίων οι παραγωγοί ακολουθούν ή είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν εξίσου αυστηρές διατάξεις για την παραγωγή τους όπως αυτές που ακολουθούν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί, ο Ούγγρος παραγωγός. Το σύστημα δηλαδή του cross compliance θα έπρεπε να ισχύει εδώ, της αμοιβαίας δηλαδή εφαρμογής των κανόνων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μόνο με απόλυτη απόδειξη το, της στήρησης των συνθήκων παραγωγής και, ευημερίας, και προστασίας ευημερίας των ζώων θα μπορούσαν να εισάγονται τα προϊόντα αυτά. Παρ' όλα αυτά, Είναι πολύ θετική εξέλιξη ότι επιβαρέται η σήμανση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και ότι εισάγεται η αρχή της ασφάλειας των τροφίμων ως προτεραιότητα μέσα από την νομοθεσία αυτή. Μπορούμε έτσι πιστεύω να προστατέψουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών και να διαφυλάξουμε και τους γεωργούς μας ώστε να υπάρχουν επαρκείς όροι ε, ισότιμου ανταγωνισμού. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μορβάη. Για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Γκροστέτ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σήμερα συζητάμε για ένα κανονισμό πολύ σημαντικό γιατί αφορά νέα τρόφιμα και η τεχνολογική καινοτομία φυσικά είναι πολύ σημαντική στο επιστημιστικό τομέα και αυτό θα πρέπει να εξυπηρετεί τον καταναλωτή και όχι να είναι του. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ε, το, το ότι κάποια από αυτά τα νέα προϊόντα είναι πιο ασφαλή. Ε, φυσικά είμαστε ε, πολύ προσεκτικοί απέναντι σε τρόφιμα από ζώα και τους απογόνους τους. Α, δεν μπορώ να δεχτώ αυτούς που λένε ότι πρέπει να υπάρχει συστηματική απαγόρευση. Ε, είναι, θα ήταν κρίμα να προωθούμε μέσω από ιδεολογήματα θέσεις για αυτά τα τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας κάνει μια πρόταση ανεξάρτητα από την απαγόρευση ή όχι. Να μην είμαστε δημαγωγικοί για επιστημονικά θέματα, για θέματα τόσο ευαίσθητα, οποία απαιτούν ε, πολλή σκέψη. Ας μην υιοθετούμε με συστηματικό τρόπο μια στάση υπαναχώρηση ή ακόμα χειρότερα μια εκ των προτέρων ε, αρνητική στάση για ένα θέμα τόσο περίπλοκο που πρέπει να εξεταστεί ε, το, εν το βάθη. Η θέση της προφύλαξης θα πρέπει να πριτανεύει, αλλά να βασίζεται όχι σε ιδεολογήματα, αλλά σε επιστημονικά στοιχεία και στην αξιολόγηση κινδύνου. Αν υπήρχε πριν από λίγε δεκαετίε αυτή η αρχή, ε, δεν θα είχε γίνει ποτέ η πρώτη μεταμόσχευση τη καρδιά και ποτέ δεν θα είχαμε σώσει εκατοντάδε ασθενεί. Φυσικά η σύνεση μα αναγκάζει να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα για τα νανοηλικά, για ε, κλωνοποιημένου για σπέρμα ε, κλωνοποιημένων τάβρων. Αλλά τα προϊόντα τα οποία ε, προέρχονται από τέτοια βοηθή, ε, τα οποία εισάγονται από το εξωτερικό, βρίσκονται ήδη στην ευρωπαϊκή αγορά. Επομένως, ας αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουλέψει ειρηνικά, ε, ήρεμα, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ε, μεγαλύτερη ασφάλεια για τον καταναλωτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συζητήσει, να τροποποιήσει και να αποφανθεί για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Ε, για δύο λεπτά. Σνέλχαρτ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε. Στην αρχή των συζητήσεων έθεσα το ερώτημα Χρειαζόμαστε νέα οδηγία, νέο κανονισμό για την ασφάλεια των τροφίμων. Δεν έχουμε αρκετή νομοθεσία. Ναι, τη χρειαζόμαστε πιστεύω. Κυρίως όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις προσπάθειες για την άρση του γραφειοκρατικού άχθους και γι' αυτό η δεύτερη ανάγνωση έχει ιδιαίτερη σημασία. Ένα τέτοιο κανονισμό για τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να ασχολείται μόνο με τα νέα τρόφιμα. Η η συγγήτρια πάντως βλέπουμε ότι εισάγει και στη δεύτερη ανάγνωση όλες τις τροπολογίες της πρώτης ανάγνωσης, ακόμη και γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει ήδη ογκοδέστατη νομοθεσία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι του οποίου προσπαθεί να εξυπηρετήσει, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει αυτό να γίνει μέσα από την επαναφορά ε, τροπολογιών από την πρώτη ανάγνωση. Επίσης, ως προς την ανοτεχνολογία. Έχουμε μια νέα εξέλιξη, μια νέα διαδικασία, αλλά ας προσέξουμε να μην παραλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος, να μην ε, κατηγορούμε για πάνω δεινό αυτή τη νέα τεχνολογία, την άνοτεχνολογία. Δεν είναι δεδομένο ότι είναι υπέτεια για τα πάντα. Έχω ενημερωθεί αρκετά για την ανατεχνολογία από τους ειδικού και βλέπω ότι προσφέρει τεράστιες δυνατότητες και γι' αυτό καλό θα ήταν να προσκαλέσουμε τους ειδικού στην Επιτροπή μας. Και Πιστεύω ότι τότε θα ομολογήσουμε όλοι ότι πρέπει να συνεχίσουμε και την έρευνα, βεβαίω όπω οφείλουμε για την ανατεχνολογία, αλλά και να επιτρέψουμε τη χρήση της και την αξιοποίησή της εκεί όπου είναι χρήσιμη. Για την κλωνοποίηση των ζώων, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια τροπολογία η οποία έχει να κάνει με την υποχρεωτική ε, δυνάμη της Συνθήκης Λισαβόνας προστασία της εφημερίας των ζώων και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο Επίτροπος έχει δεσμευθεί να καταθέσει νέο έγγραφο για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Σνέλχαρτ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Αντορέσκου. Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο στόχο της εξέτασης αυτού του κανονισμού είναι η επίτευξη ε, υψηλού επίπεδου προστασία ε, των καταναλωτών, ε, των, των ζώων και του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή τη προφύλαξης. Υπάρχουν όμω σημαντικέ αμφιβολίε όσον αφορά την ασφάλεια του κρέατο που προέρχεται από κλεινοποιημένα ζώα. Τα ζώα αυτά ε, υποφέρουν από πρόωρη γύρανση και από άλλε ασθένειε και δεν ε, είναι ξεκάθαρο στου επιστήμονε ε, οι διαφορέ όσον αφορά την υγεία των ζώων αυτών από τα υπόλοιπα. Οι περισσότεροι κλωνοποιημένοι οργανισμοί πάντω δεν επιβιώνουν επιμακρών ε, ε, ή πεθαίνουν πρόωρα. Ένα στα 75 ζώα επιβιώνει. Ε, και υπάρχουν και, και, και αμφιβολίε όσον αφορά την ασφάλεια τη τεχνική αυτή, η οποία φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για, για ανθρώπινη χρήση. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρέ ανησυχίε και απειλέ για την υγεία. Ε, και, άλλε, επιπτώσει ε, άλλες επιπτώσεις όσον αφορά τη χρήση αυτή τη τεχνική. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να είναι ξεκάθαρο. Λαμβάνοντα υπόψη επίσης τις ε, ανησυχίες, τις σωστές συνθήκες διαβίωσης ε, των ζώων, νομίζω θα πρέπει να επιμείνουμε και να απαγορεύσουμε την κλωνοποίηση και τη χρήση των κλωνοποιημένων ζώων. Ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό τώρα το λόγο και ο κύριο Φιέλνερ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συναδελφοί, Κύριε Πρόεδρε, αυτό που βλέπω εγώ στο πιάτο μου όταν κάθομαι στο τραπέζι δεν είναι το ίδιο με αυτό που έβλεπαν οι γονεί μου. Αλλά και εκείνοι είχαν άλλο φαγητό στο πιάτο τους σε σχέση με εκείνο που έβλεπαν οι δικοί τους γονείς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε να θρέφουμε τον πλανήτη. Και γι' αυτό αυτό που θα τρώνε τα παιδιά μου σε μια δεκαετία, δύο, δεν θα είναι το ίδιο με αυτό που τρώω εγώ τώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να απαγορεύσουμε νέα τρόφιμα και να τα καταδικάσουμε συλλήβδιν. Ωστόσο πρέπει να τηρούνται απαράλλακτα απαρέγκλητα τρεις βασικές αρχές. Πρέπει να στηρίζεται η νομοθεσία σε, η αδειοδότηση δηλαδή, σε επιστημονικά δεδομένα και έρευνα. Δεν πρέπει δηλαδή να τίθεται ζήτημα προσωπικής επιλογής ή προτίμησης ή ιδιαίτερων συμφερόντων. Πρέπει δηλαδή να ε, καλωσορίσουμε τις νέες εξήλιξεις και όχι να τις καταδικάσουμε εκ προημίου. Δεύτερον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι είναι ασφαλή τα νέα αυτά τρόφιμα για τον καταναλωτή, γιατί διαφορετικά ο καταναλωτής θα τα αγνοήσει, δεν θα τα προτιμήσει, δεν θα τα αγοράσει. Τρίτον, και για να κλείσω, πρέπει να βεβαιωθούμε, να βεβαιωνόμαστε σε κάθε περίπτωση ότι τα ε, συστήματα αδειοδότηση αυτών των νέων τροφίμων δεν θα αποτελέσουν νέου τελωνιακού ή μη μάλλον μη τελωνιακού φραγμού για να εμποδιστεί δηλαδή είσοδο στην αγορά των προϊόντων αυτών. Ευχαριστώ κύριε Φιέλνερ. Ε, περνάμε στην επόμενη παρέμβαση για 1,5 λεπτό τη κυρία Κλά. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, κύριε Επίτροπε, υπάρχουν νέα τρόφιμα, άρα χρειαζόμαστε νέους κανόνες, νέες ρυθμίσεις. Εδώ λαμβάνονται υπόψη και οι δεοντολογικές επιφυλάξεις προς την διάθεση στην αγορά τέτοιου είδους νέων τροφίμων, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Όπως προέκυψε και από τη σημερινή συζήτηση, καταρχάς θέτει το ζήτημα της κατανάλωσης κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα. Υπάρχει επαρκής παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρέατος που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ε, καταφύγουμε σε κρέας από κλωνοποιημένα ζώα χωρίς να είναι δεδομένο ότι επιβαρύνει την δημόσια υγεία αυτό το κρέας, ε, θα πρέπει να αποκλειστεί όσο δεν είναι γνωστό τι είδους ε, επιπτώσεις μπορεί να έχει και τι είδους ε, προβλήματα προξενεί η παραγωγή του στα ίδια τα ζώα. Γιατί είναι άγνωστο μεν το πόσο υποφέρουν τα ζώα αυτά, είναι γνωστό όμως ότι έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό επιβίωσης και χαμηλά επίπεδα υγείας δεν μπορούμε να, εισάγουμε, να εισαγάγουμε κλωνοποιημένα ζώα στην τροφική αλυσίδα και πρέπει να αποστείλουμε σαφές πολιτικό μήνυμα και στην Επιτροπή όπως και στον πολίτη. Ένα άλλο ζήτημα αυτού του κανονισμού είναι η ρύθμιση σχετική με την ανοτεχνολογία για να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο για προστασία του καταναλωτή, του τελικού χρήστη δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας οριζόντιος ε, ορισμός που θα ισχύει απανταχού όχι μόνο για τα νέα μέσα, για τα νέα τρόφιμα αλλά και για την, που θα καλύπτει και την οδηγία για κάθε είδος προϊόντος ε, καλοπισμού ε, ή αντίστοιχου που έρχεται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα και τον ανθρώπινο οργανισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροντσούλη τώρα για να κλείσει η συζήτηση. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οχτώ Ευρωπαίοι στους δέκα θεωρούν ότι δεν είναι δικαιολογημένη η κλωνοποίηση των ζώων για διατροφικούς λόγους και έξι στους δέκα δηλώνουν ότι αποκλείεται να καταναλώσουν τέτοια προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα. Αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ακόμα μια φορά ότι δεν υπάρχει λόγος να κλωνοποιούμε τα ζώα για διατροφικούς λόγους. Το να επιτρέψουμε την εμπορία τροφίμων που παράγονται από κλωνοποιημένα ζώα ε, θα πρέπει να μας κάνει όλους να σκεφτούμε για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας επιλογής. Το να επιτρέψουμε την κατανάλωση ε, τρο, κρέατος, γάλακτος και τυριών από τέτοια ζώα μπορεί να οδηγήσει σε προϊόντα τα οποία δεν είναι υγιή και που δημιουργούνται τεχνητά μέσα στα εργαστήρια. Όπω είπε και η κυρία Αντωνέσκου, δεν ξέρουμε αν η κλινοποίηση για διατροφικό λόγο είναι ασφαλή και δεν περιέχει ε, κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Ξέρουμε ότι απλώ η τεχνολογία αυτή προκαλεί φοβερό πόνο και αρρώστια στα ζώα αυτά. Τα τρόφιμα αυτά επίσης ε, θέτουν αμφιβόλο την ε, παραγωγή των κλασικών προϊόντων και χιλιάδων ε, εκμεταλλεύσεων που με φοβερές θυσίες εξασφαλίζουν προϊόντα αριστείας κάθε μέρα. Επομένως δεν θέλουμε τέτοια προϊόντα στα τραπέζια μας. Θέλουμε μια διατροφή υγι... υγιεινή, ασφαλή και μεσογειακή δυνατόν. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ε, τελειώσαμε λοιπόν με τις παρεμβάσεις ε, και περνάμε τώρα ε, στο τμήμα Catch the Eye. Ξέρετε ότι ο κανόνας είναι να δίνουμε το λόγο σε πέντε συναδέλφους. Εφτά συνάδελφοι όμως που έχουν ζητήσει το λόγο. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο και στους εφτά. Αλλά να ξέρετε ότι μόλις τελειώσει το λεπτό θα σας διακόπτω. Πρώτα απ' όλα η κυρία Κόστιγκερ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγητριά για τη δουλειά της. Είναι πολύ θετικό το ότι επιτέλους με αυτή τη για το νέο κανονισμό και τα νέα τρόφιμα μπορούμε να έχουμε γενικές διατάξεις που θα ρυθμίσουν τη διάθεση των τροφίμων αυτών στην ευρωπαϊκή αγορά με ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή. Έχουμε να κάνουμε πάνω απ' όλα με διοντολογικές αλλά και με υγειονομικές πτυχές που σχετίζονται με την κατανάλωση κρέατος αποκλωνοποιημένα ζώα. Απαιτείται ύψιστη ύψιστο επίπεδο προστασία του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ανεξαρτήτως του τρόπου παραγωγή. Θέλουμε να έχουμε τι καλύτερε συνθήκε παραγωγή στη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα όσον αφορά τα τρόφιμα που απευθύνονται στην ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να έχουμε τι αυστηρότερες προποθέσει προστασία και πρόληψης. Γι' αυτό δεν πρέπει να καταναλώνουμε κρέα από κλωνοποιημένα ζώα. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος διακόψε την ομιλήτρια. Ευχαριστώ η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και απευθύνω παράκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη τα όσα υπόθηκαν σήμερα. Χρειαζόμαστε νέο κανονισμό για τα νέα τρόφιμα που θα διατίθενται στην αγορά κατά τρόπο ασφαλή. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι κλωνοποιημένο κρέας. Χρειαζόμαστε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν χρειαζόμαστε αυτοκλωνοποιημένο κρέας. Οι καταναλωτές, οι Ευρωπαίοι έχουν απορρίψει τα προϊόντα αυτά και νομίζω ότι εάν ε, αληθεύει το ότι το να απορρίπτονται τα προϊόντα αυτά ως επικίνδυνα δεν είναι επιστημονικά βάσιμο, ταυτόχρονα δεν μπορούν αυτά τα προϊόντα και να διατίθεται στις αγορές πριν βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για την υγεία του καταναλωτή. Κάθε είδους αμφιβολία θα πρέπει πρώτα να έχει διασκεδαστεί και μετά να διατεθούν τα, τα, προϊόντα αυτά στην αγορά. Αυτά προς όφελος και του καταναλωτή αλλά και της γεωργίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην χρήση των ανοηλικών στα τρόφιμα. Πράγμα το οποίο γεννά πολλές ανησυχίες και αμφιβολίες για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Ήδη διατυπώνονται πολλέ επιφυλάξει, διότι δεν είναι ικανοποιητικέ οι επιστημονικέ γνώσει που έχει συλλέξει η επιστημονική κοινότητα ω προ τι συνέπειε τη χρήση νανοηλικών στα τρόφιμα και ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αυτά συμπεριφέρονται μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αυτό δεν πρέπει επουδενή να επιτραπεί η χρήση τέτοιων υλικών στα τρόφιμα πριν γίνουν πληρέστατε μελέτε και έρευνε για τι συνέπειέ του ω προ τη δημόσια υγεία και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να εκφράσω τον βαθύτατο θαυμασμό, θαυμασμό μου για την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος και έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Ντάλι, θα ήθελα να μιλήσω για την απαγόρευση των, της θέσης στην αγορά α, προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα και από γόνων τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ε, δεν υπάρχει ε, υπάρχουν, υπάρχει ποσότητα κρέατος στην ευρωπαϊκή αγορά και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να καταφύγουμε σε τέτοιο κρέας που δημιουργεί και διοντολογικά προβλήματα. Ε, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ομάδα Διοντολογίας ε, και θα ήθελα να σας μιλήσω για τα επιστημονικά πορίσματα που υπάρχουν για την υγεία των ζώων, το περιβάλλον. Υπάρχουν ελλειπείς γνώσεις ε, για τα κλωνοποιημένα ζώα, τους απογόνους τους. Αυτή η ομάδα διοντολογίας δεν θεωρεί ότι υπάρχουν πιστικά επιχειρήματα για να θέσουμε στην αγορά, κόβεται ο μιλητής, ο κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Επίτροπε, το θέμα της απαγόρευσης κλωνοποιημένων ειδών στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ένα θέμα πραγματικά σεβασμού της αρχής της πρόληψης όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή συνθήκη στη συνθήκη λισαβόνας στο άρθρο. 191. δεν έχουμε επαρκείς ε, μελέτες ούτε για τις ε, επιπτώσεις στην υγεία ούτε για τις επιπτώσεις στην, ε, στα ζώα από την, χρήση των, την παραγωγή κλωνοποιημένων ειδών. το ίδιο ισχύει για τις νανοτεχνολογίες ενώ ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε αυτή την οδηγία είναι η σήμανση των μεταλλαγμένων προϊόντων αν οι ευρωπαίοι πολίτες έχουμε δικαίωμα να επιλέγουμε αν θα καταναλώνουμε ή όχι μεταλλαγμένα προϊόντα τότε θα πρέπει να έχουμε και τη γνώση αν ένα προϊόν ε, έχει καταναλώσει ή είναι προϊόν επεξεργασίας ε, και παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν μεταλλαγμένα ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το λόγο έχει η κυρία Ντότζ. Ε, Επίτροπε, πιστεύω ότι τα κλωνοποιημένα ζώα ε, ή οποιοδήποτε προϊόν που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να εξετάσει δεόντως ε, το πώ θα αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό και στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα κανένα προϊόν που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα ή του απογόνους του δεν θα πρέπει να υπησέρχεται στην τροφική άλυσο. Η νέα τεχνολογία χρησιμοποιείται ευρέω σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε ε, ε, προϊόντα τα οποία όμως, για τα οποία όμω θα μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ακολουθείτε διαφάνεια σε ολόκληρη τη διαδικασία ε, ε, παρασκευής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη πιστοποίηση, έγκριση, έλεγχο και ετικετοθεσία με τρόπο που να μην παραπλανά τον καταναλωτή. Ε, και τα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτε χώρε θα πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ισχύουν για τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πληρούνται όλε οι προποθέσει. Διακόπτεται ε, το λόγο έχει τώρα η κυρία Ροϊτόβα, λέει ο πρόεδρος. Ε, Ευχαριστώ. Ως εισηγήτρια για την γνωμοδότηση στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στη δεύτερη ανάγνωση. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη θέση στην αγορά, ε, μεγαλύτερη ευκολία για τη θέση στην αγορά, ε, μεγαλύτερη ασφάλεια. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Διοντολογίας πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης, ε, υπάρχει ένα πρόβλημα με, το, με τα τρόφιμα που εμπεριέχουν γάματα φόμικρον. Είναι αντικείμενο μιας άλλη οδηγία βέβαια αυτό και θα πρέπει να ζητήσουμε την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Το Κοινοβούλιο επίσης θα πρέπει να ζητήσει το κρέα από κλωνοποιημένα ζώα να μην συμπεριληφθεί. Τελειώνουμε τον κύριο Σιλβέστρης. Θα πρέπει να επιτρέψουμε την εμπορευματοποίηση κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα, ε, λέει. Γιατί Έχουμε έλλειψη σε κρέα στην Ευρώπη σε καμία περίπτωση. Δεν στέκει αυτό το επιχείρημα. Δεν υπάρχει επαρκή πληροφόρηση στους καταναλωτές. Μπορεί ο καταναλωτής ε, να καταλάβει ε, ποιο κρέας προέρχεται από ποιο ζώο και ποιο κρέας προέρχεται από κλωνοποιημένο ζώο. Δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες, δεν έχουμε καθόλου στοιχεία για τη διατροφική αξία των ε, προϊόντων αυτών. Ε, ίσως χρειαζόμαστε ακόμα 50 χρόνια για να καταλάβουμε κάποια πράγματα για αυτά τα νέα τρόφιμα. Ε, κάθε φορά που υπάρχει μία επιδημία, ε, περιμένουμε χρόνια και χρόνια για να καταλάβουμε την αιτία αυτών των επιδημιών. Τώρα βάζουμε νέα δηλαδή τρόφιμα στην αγορά όταν δεν υπάρχει επιστημονική ασφάλεια. Ε, η Ευρώπη δεν θέλει να ξέρει από πού προέρχονται αυτά τα προϊόντα. Διακόπτεται ο μιλητής. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Και τελειώνουμε αυτό το γύρο με τον Επίτροπο Ντάλι. Θα απαντήσει στα διάφορα ερωτήματα και στις διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν. Κύριε Ντάλι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να υποστηρίξω τις εξής αρχές. Καταρχάς, η αποκεντρωπημένη διαδικασία ε, αντικαθίσταται με μια συγκεντρωτική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, η απόφαση για την αδειοδότηση λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια διαδικασία με βάση κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές για τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, ούτω ώστε να έχουμε ασφαλή τρόφιμα τα οποία ε, υπόκειται σε διαδικασίε ε, ελέγχου και διαχείριση του κινδύνου. Για να υπάρξει καινοτομία και ασφάλεια στα τρόφιμα, θα πρέπει ε, να δούμε τι γίνεται με την προστασία των δεδομένων για τα νέα τρόφιμα. Επίσης, θα πρέπει να ορίσουμε με επιστημονικό τρόπο τα νανοηλικά, τα οποία, ο οποίος ορισμός θα, θα προσαρμόζεται ανάλογα στην εξε, με τις εξελίξεις της επιστήμης. Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από τους πολιτικούς, αλλά από τους επιστήμονες. Πέμπτον, διευκρίνηση του γεγονότος ότι όλα τα τρόφιμα τα οποία έχουν νανοηλικά θα πρέπει να εξετάζονται και να διοδοτούνται ανά περίπτωση και έκτον το δικαίωμα των καταναλωτών να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει συστηματική ετικετοθεσία όλων των προϊόντων που έχουν ανοηλικά. Σε ό,τι αφορά την κλωνοποίηση, άκουσα τι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα εξετάσω πολύ προσεκτικά αν η νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα είναι το κατάλληλο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τα κλωνοποιημένα ζώα και τα προϊόντα από τέτοια ζώα γιατί αυτό το θέμα ξεπερνάει το εύρο και το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Κυρία Γκροστέτ, σας διαβεβαιώ ότι η έκθεση για την κλωνοποίηση θα την επεξεργαστούμε με ψυχραιμία και θα λάβουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία ε, των τροφίμων που παράγονται από κλωνοποιημένα ζώα και από γόνους τους και περιμένουμε να γίνει μια ενδελεχή συζήτηση με το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Ο στόχος είναι η έκθεση αυτή να οδηγήσει σε ισορροπημένε λύσεις, ούτω ώστε να διασκεδαστούν όλες οι ανησυχίες όλων των θεσμικών οργάνων με βάση τι τις θεσμικές υποχρεώσεις και τις του υποχρεώσεις. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Τελειώνει λοιπόν η συζήτηση με την παρέμβαση για δύο λεπτά της εισηγήτριας, της κυρίας Λίοταρτ. Σας ευχαριστώ και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους ε, εσάς που συμμετείχατε με τόσο ενδιαφέρον συζήτηση. Βεβαίως λυπούμε ε, που λάβει για τις απουσίες του το Συμβούλιο, διότι πιστεύω ότι θα ήταν επιθυμητό και το Συμβούλιο να μπορέσει να ακούσει τη σαφή μας τοποθέτηση. Και λυπάμαι ε, ακριβώς διότι Ε, δεν γίνεται δημόσια συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Προσωπικά πρέπει να σας πω ότι δεν ε, ε, θέλω να, βρε, βρω στο πιάτο μου κλωνοποιημένα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει σαφή νομοθεσία και θα πρέπει να πούμε ότι απαιτείται ξεχωριστή νομοθεσία και δεν πρόκειται μέσα από, τα, από τη νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα να λύσουμε το ζήτημα του κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα. Το ίδιο ισχύει και για την ανατεχνολογία η τεχνολογία ε, και ε, τα κλωνοποιημένα ζώα συζητούνται πολύ ε, επιμακρών. Αλλά εδώ μιλάμε, δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα σημεία, μιλάμε και για την τεχνολογία που βρίσκεται στο στάδιο της ανακάλυψης ή για τις προσεχείς ανακαλύψεις της τεχνολογίας. Και βεβαίως δεν θέλουμε να παραβλέψουμε τις ανακαλύψεις αυτές. Απλά και μόνο θέλουμε να ξέρει ακριβώς τι καταναλώνει ο καταναλωτής. Και θα πρέπει ε, να είμαστε σίγουροι ότι προσφέρουμε ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή. Αυτή η συζήτηση λοιπόν για την κλωνοποίηση ελπίζω να μην αποτελέσει εμπόδιο για την ε, έγκριση της νομοθεσίας για τα νέα τρόφιμα. Γιατί πράγματι υπάρχουν αρκετές χώρες που ε, ε, αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Τρίτες χώρες που θέλουν τα παραδοσιακά τους τρόφιμα να τα εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς τους δημιουργούμε εμπόδια. Μα δεν υπάρχει λόγος. Όταν πρόκειται για φυσικά τρόφιμα, αν θέλετε, για τρόφιμα που προέρχονται από τη φυσική οδό, δεν υπάρχει λόγος μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Ε, λυπάμαι λοιπόν που το Συμβούλιο δεν είναι σήμερα εδώ. Ελπίζω πάντω ε, το θέμα να λυθεί ευνοϊκά. Σα ευχαριστούμε για την παρέμβασή σα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι μάλλον. Αύριο στι 12 η ώρα. Λοιπόν, το επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Κράμερ για τις βιομηχανικές εκπομπές, ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρήπανσης. Αναδιατύπωση.